Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε την κοινή συζήτηση για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας. Έχουμε τη σύσταση Σβόμποντα για τη συνθήκη προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας και στην έκθεση πάντα του κυρίου Χάνες Σβόμποντα για την αίτηση της Κροατίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσω το λόγο αμέσως στον ομιλητή για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε από το Συμβουλίο, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί επισκέπτε από την Κροατία με τα επικεφαλή του Λουκα τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τον κύριο Διαπραγματευτή και ε, πρέσβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ομολογώ, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι είμαι συγκινημένο και ευτυχή που μπορώ να υποβάλω στο Κοινοβούλιο σήμερα τελευταία μου έκθεση για την Κροατία και να ζητήσω να συμφωνήσετε με την προσχώρηση τη Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μακρά και δύσκολη η διαδικασία αυτή και κατά τη διάρκεια αυτή τη διαπραγμάτευση είχα να κάνω με τη Μεσοράτσα, τον και τον Φεδρικόσο, τρει πρωθυπουργού και πολλού άλλου πολιτικού Βεσναπούζη, ο Μιλάνοβιτ και Μίλοβατ Πόποβατ. Όλοι οι πολιτικοί αυτοί πέρα από τα κομματικά όρια δείχθηκαν ανοιχτοί και αναγνώρισαν ότι θα πρέπει από κοινού να κινηθούν στα ευρωπαϊκά θέματα. Αυτό είναι καλό παράδειγμα και για τις άλλες χώρες της περιοχής. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις εισηγητές. Συνεργαστήκαν πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την Εκτελεστική Επιτροφή και τον Επίτροπο Φίλε ιδιαίτερα. Και αν είναι δυνατόν ευχαριστήσω και το Συμβούλιο. Μόνο μία συνεπής πολιτική από την ευρωπαϊκή πλευρά μας επέτρεψε μαζί με τους υπεύθυνους πολιτικούς Κροατίας να πετύχουμε η Κροατία να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και κυρίως τη συνεργασία με το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και δεν είναι θέμα εκδίκησης, δεν είναι θέμα ευαισθησιών ευρωπαϊκών, αλλά θέμα αντιμετώπισης της ίδιας της ιστορίας και της επεξεργασίας των σφαλμάτων του παρελθόντος. Εγώ δεν το ενώνησα ποτέ ε, σαν μια κριτική προς την Κροατία, αλλά μια κριτική ότι κατά πάσα πιθανότητα ορισμένοι εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση για να παράξουν εγκλήματα πολέμου. Επίσης πολλά γίνουν όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και το γεγονός ότι ένας τέος πρωθυπουργός ε, είναι αυτή τη στιγμή ενώπιον δικαστηρίου δεν αποδεικνύει ότι υπάρχει πολλή διαφθορά αλλά ότι στην Κροατία αντιμετωπίζουν το θέμα της ε, διαφθοράς και το καταπολεμών. Και έγιναν πολλά σημαντικά βήματα όσον αφορά την ε, μεταρρύθμιση δικαιοσύνης και θα υπάρχει μια επιτήρηση που είναι κατά τη γνώμη μου σημαντική γιατί θα πρέπει η Κομισιόν να φροντίσει πριν από την πραγματική ένταξη να προωθηθούν οι ε, μεταρρυθμίσεις. Επίσης πολλά έγιναν για την ενσωμάτωση στην κοινωνία αυτή των Σέρβων που παλινώστησαν και είναι καλό να υπάρχουν κοινά βήματα, ας πούμε όπως με την επίσκεψη αυτή στην Βούκοβα. Λίγες εβδομάδες μετά τη φρικτή καταστροφή πήγα εγώ στην Βίκοβα και είδα τι μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα επιθετική στάση που ε, δαυλίζεται και από πολιτικούς. Από την άλλη μεριά είδα ότι στη Βούκοβα ζουν πολλοί που έχουν κατά νου το μέλλον και είδα με ένα κοινό σχολείο κρατών και Σέρβων και είδα πώς προτίθεται να συζητήσουν για το μέλλον. Είχα μία από τις καλύτερες συζητήσεις ποτά και ε, στην Βούκοβα ήξεραν περί τίνος πρόκειται στην Ευρώπη που πολλοί από εμάς δεν το ξέρουν. Να ξεπεράσουμε δηλαδή τα μίση και τις διαμάχες. Και είδα ότι το ποτάμι εκεί όσο πάει και ενώνουν τους ανθρώπους και δεν τους χωρίζει. Και αυτό είναι σημαντικό. Θα ήθελα να προσθέσω δύο λεπτά κύριε Πρόεδρε. Και επίση είπα ότι είμαι ότι ακριβώ λόγω αυτών των σκέψεων, η Κροατία θα κάνει ό,τι χρειάζεται, ούτω ώστε να δώσει στι άλλε χώρε τη περιοχή την δυνατότητα προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική τη είναι πολύ σημαντικό τομέα και ήθελα να επαναλάβω ότι είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που και η Κροατία και η Σλοβατία και ήθελα να αναφέρω εδώ τον ε, Δήμαρχο Ποτάχα της ε, στη χώρα αυτή που κατάφερε να καταβάλει προς πολλές προσπάθειες να ξεπεραστούν οι διαμάχες στα σύνορα. Το παράδειγμα της ε, Κροατίας είναι για μένα ένα σημαντικό βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ελπίζω να είναι τολμηρό αρκετά το Συμβούλιο ούτω ώστε τις επόμενες μέρες να κάνει ένα βήμα στον αφορά τη Σερβία και το Μαυροβούνι ούτω ώστε να προωθηθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης και μετά την ένταξη Κροατίας. Ξέρω ότι πολλοί σκέφτονται μήπως θα έπρεπε ε, να δούμε τι γίνεται με τα, με σημερινά μας προβλήματα και κατά πόσον αυτές οι συνεχείς προσχωρήσεις δεν οδηγούν σε περισσότερα προβλήματα. Όχι, όχι. Δεν ε, έφταιγαν οι νέες χώρες για τα προβλήματά μας. Και ελπίζω αύριο να υπάρχει ευρεία συνένεση για την ένταξη της δυσκολίας και να δοθεί έτσι ένα πνεύμα ελπίδας, εμπιστοσύνης, ιδίως εν ώψη τους, ε, της μερολατρίας και της απεσιοδοξίας που υπάρχει. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε με την κροματεία μαζί να προχωρήσουμε, να προωθήσουμε την Ευρώπη δίνοντας ένα μήνυμα ότι πραγματικά πιστεύουμε σε αυτή την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Πολύ πήρατε και τον χρόνο της δευτερολογίας. Τώρα ερχόμαστε στον ε, Υπουργό, τον κύριο Ντογγέλεβιτς, εξ ονόματος του Συμβουλίου. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητά μέλη, <clears throat> σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να πάρω μέρος στη συζήτηση αυτή Είμαστε στα τελικά βήματα της διαδικασίας που θα οδηγήσει σε λίγες μέρες στην υπογραφή της Συμφωνίας Ένταξης, της Συνθήκης Ένταξης, που θα οδηγήσει στη δημιουργία του 28ου κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτους μέλους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει να συγχαρώ την Κροατία, η οποία πέτυχε να ολοκληρώσει με επιτυχία θα έλεγα την ε, μακρόχρονη αυτή προενταξιακή περίοδο. Νομίζω ότι η πολιτική διεύρυνση είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει σαν βασικό στόχο την ενίσχυση της ειρήνης και την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Και η διεύρυνση είναι ο βασικός τρόπος για να τα πετύχουμε αυτά. Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τα προβλήματα που συζητούσαμε πριν λίγο, η ένταξη μας υπενθυμίζει γιατί οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν να ολοκληρωθούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πετύχει η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και πολλές χώρες θέλουν να γίνουν κομμάτι αυτής της επιτυχίας. Το κοινοβούλιο αυτό, χωρίς καμία διακοπή, στήριξε τη διαδικασία ένταξης και θέλω να το ευχαριστήσω για αυτή του την υποστήριξη. Να υπογραμμίσω επίσης ότι βασική βασικός θα έλεγα θεμέλιο της ομοφωνίας για τη διεύρυνση είναι η εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων τις οποίες θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι απαραίτητες για να γίνει κανείς μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να γίνει κανείς μέλος της Ένωσης ε, φέρει κάποια πλεονεκτήματα, αλλά ταυτόχρονα και αρκετές υποχρεώσεις, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν πλήρως τη διαδικασία ένταξης και την ίδια την ένταξη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να υπογραμμίσω ιδιαίτερα. Υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό κομμάτι θα έλεγα στον τομέα της αξιοπιστίας αν η υποψήφια χώρα εκπληρεί τις προϋποθέσεις, θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τις δικές της υποσχέσεις. Εφόσον συμφωνήσετε λοιπόν κι εσείς για την ένταξη, θα μπορέσουμε να την υπογράψουμε σύντομα εδώ στις Βρυξέλλες. Η Πρωθυπουργό της Κροατίας, η κυρία Κόσορ, θα μπορέσει να πάρει μέρος σαν παρατηρήτρια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το απόγευμα της ίδιας μέρας είναι μια νότα αισιοδοξία και μια νότα θα έλεγα ενωτική για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Να αναφερθώ επίσης ότι η εργασία για την ένταξη της χώρας αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Η Κροατία, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ιουνίου, θα συνεχίσει τις προσπάθειές της έτσι ώστε να μπορέσει να τηρήσει πλήρως τις ανηλυμένες της υποχρεώσεις και περιμένουμε λοιπόν περαιτέρω ε, θα έλεγα βελτιώσεις. Η στενή εποπτεία θα συνεχιστεί και αυτή, ιδιαίτερα στα θέματα σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της μεταρρύθμισης στον τομέα της δικαιοσύνης και των δημοσίων ελευθεριών. Το Συμβούλιο εξέτασε προσεκτικά τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, Κροατία και τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις της τελευταίας φάσης για τα διάφορα κεφάλαια. Θα συνεχίσουμε λοιπόν εμείς να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα σας πληροφορήσουμε δεόντως και δεν μην ξεχνάμε το μέλλον. Η ένταξη της Κροατίας έχει μεγάλη σημασία για το σύνολο της περιοχής. Είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα και σαν τέτοιο θα πρέπει να αναγνωστεί έτσι ώστε να ενισχυθεί η ειρήνη, η συμφιλίωση, η ελευθερία και η δημοκρατία και οι σωστές γειτονικές και ειρηνικές γειτονικές σχέσεις, σχέσεις ανάμεσα σε γείτονες. Θα είναι, θα έλεγα, η ένταξη της Κροατίας ε, μια ενθάρρυνση για τις υπόλοιπες χώρες να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία που ακολούθησε η Κροατία, να συμφιλειωθούν με τους γείτονές τους, και να αποδείξουν την αποφασιστικότητά τους να εκπληρούν και αυτές τα κριτήρια ένταξης. Η τελετή της 9ης Δεκεμβρίου θα δώσει μια νέα όθηση για την πρόοδο και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων, εφόσον βέβαια όλες οι χώρες εμείνουν στις προσπάθειες τις οποίες κάνουν πολύ κύριε Υπουργέ. Τώρα θα πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι από τις ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ο κύριος Φάρμ πρώτα για ένα λεπτό από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Παρακαλώ κύριε συνάδελφε. με ε, I apologize. Κύριε Επίτροπε, σας ζητώ συγγνώμη. συγγνώμη. Πρώτα ο κύριος Φίλε. Κύριος Επίτροπος έχει το λόγο πρώτα. Συγγνώμη. Ναι, Δεν πειράζει κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, έντοιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα είναι μια αποφασιστική καμπή στην πορεία της Κροατίας να γίνει το 28ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλείστε εσείς να δώσετε την έγκρισή σας. Εγώ ξέρω ότι σήμερα είναι πολλοί Κροάτες οι οποίοι εργάστηκαν πάρα πολλά χρόνια για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Κυρία Πρόεδρε, η Κομισιόν έχει ήδη δώσει τη θετική της γνωμοδότηση στις 12 Οκτωβρίου. Ελπίζω ότι η αυριανή σας ψήφος για, το, για τη σύσταση και το ψήφισμα του κυρίου Σφόμποντα θα είναι θετική. Αυτό θα επιτρέψει στο Συμβούλιο να αποφασίσει για την ένταξη της Κροατίας, ώστε η συνθήκη προσχώρησης να μπορέσει να υπογραφεί στις 9 Δεκεμβρίου. Η ψήφο σα θα είναι μια ψήφο υπέρ της Κροατίας, αλλά και υπέρ όλης της περιοχής και υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα είναι μια ψήφος υπέρ της Κροατίας. Μιας Κροατίας η οποία <clears throat> είναι πολύ διαφορετική από τη χώρα η οποία είχε σχεδόν πριν από 10 χρόνια υποβάλει μια αιτήση ένταξης. Εκεί φάνηκε η μετασχηματιστική ικανότητα της διαδικασίας ένταξης σε πολλές πτυχές της. Η οικονομία της Κροατίας είναι έτοιμη να ενταχθεί στην εσωτερική αγορά και έχει αντιμετωπίσει καλά την χρηματοπιστωτική κρίση παρά το γεγονός ότι σήμερα η Κροατία μέσα στις δύσκολες αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες μεταρρύθμισης. Πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι δημοκρατικές αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα την χάνουν σεβασμού και το κράτος δικαίου έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα από μια σειρά μεταρρυθμίσεων. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα της μεγάλης προσπάθειας και της σκληρής εργασίας της Κροατίας σε όλα τα επίπεδα. Η Κροατία είναι η πρώτη υποψήφια χώρα η οποία συνεπλήρωσε τις, ε, δια, τις ε, διαδικασίες διαπραγματεύσεων για την ένταξη με βάση της νέας μεθοδολογίας που βασίζεται σε βαθμονόμηση, σε benchmarks. Κατέδειξε η Κροατία λοιπόν ότι εκπληρεί τις αυστηρές προϋποθέσεις και επομένως θα μπορέσει να γίνει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιουλίου του 2013 υπήρξε ιδιαίτερη εστίαση στη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα και στον αγώνα κατά της διαφθοράς. <coughs> Αυτό βοήθησε ιδιαίτερα και κατήφθηνε <coughs> την Κροατία καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Οδήγησε επίσης σε αυτά και σημαντικά αποτελέσματα στην Κροατία. Παραδείγματο χάρη, ο τρόπο με τον οποίο οι δικαστικέ και ιδιοκτικέ αρχέ τη Κροατία αντιμετωπίζουν περιπτώσει διαφθορά. Δεν είναι βέβαια το τέλος της ιστορίας αυτό. Η Κροατία πρέπει να καταδείξει ότι θα σταθεί στο ύψος των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει μέσα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να συνεχίσουν οι προετοιμασίες για την ένταξη. Η περάτωση των προετοιμασιών αυτών θα είναι ένας σημαντικός στόχος για την κυβέρνηση που θα προέλθει από τις εκλογές του Δεκεμβρίου στην Κροατία. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει την παρακολούθηση και τις εκθέσεις της για τον σεβασμό από την πλευρά της Κροατίας των υπεσχημένων, των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει, με τρόπο ο οποίος θα είναι ενδελεχής και αντικειμενικός. Μέχρι τη στιγμή της ένταξης λοιπόν θα συνεχίσουμε και να βοηθούμε την Κροατία σε αυτό το τελικό στάδιο προετοιμασίας. Η Κομισιόν θέλει επίση να συνεχίσει να κρατεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πλήρω ενήμερο και είμαι πάντα στη διάθεσή σα για να συζητήσω τα πορίσματά μα σε σχέση με την Κροατία. Κύριε Πρόεδρε, αυτό επίσης η θετική ψήφος για την Κροατία είναι μια θετική ψήφος και για την περιοχή των Βαλκανίων, της, περιοχή, περιοχής που βρίσκεται η Κροατία. Έδειξαν ότι, έδειξε ότι και για άλλες χώρες η ένταξη είναι ένας εφικτός στόχος και ότι μπορεί να δώσει σημαντικά οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα. Είναι ο δρόμος προς την περιφερειακή συνεργασία και προς τη σταθερότητα. Είναι αυτό που καθοδηγεί την προσπάθεια επίτευξης δημοκρατικών συνθήκων και κράτους δικαίου. Είναι και ο δρόμος για να υπάρξει ανύψωση του βιωτικού επίπεδου στα κράτη αυτά που είναι υποψήφια. Δεν είναι μονάχα λοιπόν η διαδικασία ένταξης ή ευθυγράμμιση της νομοθεσίας. Είναι πάνω απ' όλα μια αλλαγή της ίδιας της κοινωνίας, μια μεταμόρφωση, μια αποδοχή των αξιών στις οποίες βασίζεται η ευθυγραμμιση της νομοθεσιας ειναι πανω από ολα μια αλλαγη Ένωση. Αυτές οι αξίες συνδέονται πάρα πολύ με τα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, της απονομής δικαιοσύνης, την ελευθερία και την ασφάλεια. Έχουμε, επομένως, δημιουργήσει μια νέα προσέγγιση. Στις προσεχείς μας διαπραγματεύσεις θα αντιμετωπίσουμε πρώτα τα θέματα αυτά και θα είναι και το τελευταίο κεφάλαιο που θα κλείνουμε. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμο μέλη του Κοινοβουλίου, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι αυτή η ψήφος είναι και μια ψήφος υπέρ της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διεύρυνση είναι προς το στρατηγικό μας συμφέρον για την ευμάρεια και την ασφάλειά μας. Η ενσωμάτωση, ο ενστερνισμός από τα Δυτικά Βαλκάνια των αξιών μας είναι ο δρόμος για μια μεταρρύθμιση η οποία είναι μη αντιστρεπτή. Η εισαγωγή τους και η ενσωμάτωσή τους στην ενιαία αγορά βοηθάει και τους εξαγωγείς μας και τους επενδυτές μας. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας σε τομείς όπως είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, το περιβάλλον και άλλα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αξιόπιστη πολιτική λοιπόν διεύρυνση είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια μας για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τη διαδικασία αυτή μεταρρύθμισης και μετασχηματισμού. Η ένταξη της Κροατίας καταδεικνύει λοιπόν ότι αυτή η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πράγματι αξιόπιστη. Θα ήθελα εν κατακλείδη να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας και για την υποστήριξή σας. Χωρίς αυτή την υποστήριξη αμφιβάλλω αν θα μπορούσαμε σήμερα να κάνουμε, να γράφουμε πια την ιστορία με αυτή την ιστορική ψήφο. Και τώρα ερχόμαστε στους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ο κύριος Φάρμ για ένα λεπτό από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, παρακαλώ. Κύριε Kroatiens medlemskap en historisk Αγαπητοί συνάδελφοι, η ένταξη της Κροατίας είναι ένα ιστορικό συμβάν. Ελπίζω και οι υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να ακολουθήσουν. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, αξιολόγησε τις οικονομικές πλευρές της ένταξης Κροατίας. Θα υπάρχει αύξηση φυσικά του κοινοτικού προϋπολογισμού και η Κροατία θα μπορέσει να βοηθήσει ακόμα περισσότερο την οικονομική ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο, η ένταξή της για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι καθοριστική. Είμαστε πεπισμένοι ότι η χώρα είναι σε θέση να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο, όπως και προσπάθησε και πέτυχε να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κροατία δεν είναι κόστος, είναι επένδυση στην οικονομική ανάπτυξη, στη δημοκρατική ανάπτυξη, στο περιβάλλον κτλ. Αυτό είναι κάτι το θετικό λοιπόν για όλη την Ευρώπη, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Καλώς όρισες Κροατία. Επί συνταγματικών υποθέσεων θα πάρει το λόγο ο κύριος Τραυσκόφσκι για ένα λεπτό επίσης. It is a η στιγμή. Κατέληξε η διαδικασία της Κροατίας, καταλή ε, η διεύρυνση αυτή για την ε, απαιτούμενη αλλαγή στην περιοχή, στην Ευρώπη και για την ανάπτυξή της. Θα ήθελα να πω ότι οι διαδικασίες για την υιοθέτηση της συνθήκης ένταξης της Δημοκρατίας της Κροατίας και τα πρωτόκολλα επίσης για την Ιρλανδία και την Τσεχία έχουν διαφορετικές νομικές βάσεις ε, το 49 και 43 και δεν μπορούν να ενταχθούν σε μία ενιαία πράξη. Μπορεί οι δύο διαδικασίες να συμπίπτουν χρονικά, να αντικατοπτρίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ήδη από τον Οκτώβριο του 2009, αλλά οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στις δύο διαδικασίες σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καθυστερήσει την ημερομηνία ένταξης της Κροατίας. Αυτό είναι απαραίτητο θα ήθελα να πω για τους φίλους μας τους Κροάτες που είναι στην τελευταία φάση της ένταξης. Καλώς ήρθατε στην Κροατική. Εξ των πολιτικών ομάδων για την ε, ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα πάρει το λόγο ο Πόσελτ. Για δύο λεπτά κύριε συνάδελφε. Frau Präsidentin. Πρόεδρε, το Σώμα υποστηρίζει την Κροατία εδώ και πάνω από 30 χρόνια σαν ε, βοηθός του Ότοφον τη ε, δεκαετία του 80 συνεργάστηκα ούτω ώστε οι πρώτοι ε, ε, πρόσφυγες Κροάτες, οι πρώτοι προσπιστές των αυτών των κομμάτων να έρθουν εδώ στο Στρασβουργό και να μας ενημερώσουν για την επιθυμία ελευθερίας του κροατικού λαού και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συμβάλαμε στην διαδικασία εκδημοκρατισμού το 1990 στις πρώτες ελεύθερες εκλογές και επί ένα χρόνο προσπαθήσαμε ό,τι μπορούμε για να επιστήσουμε την προσοχή των κρατών ότι χρειάζεται να υπάρχει διαπραγμάτευση με το Βελιγράδι για μια ειρηνική μετατροπή της ε, Ιουγκοσλαβίας σε μια ε, ένωση κρατών στην οποία θα ανήκει και η Κροατία. Αυτά απέτυχαν όμως γιατί πολλοί στην δυτικό κόσμο κοιμόντουσαν και επίσης ήταν άκαμπτοι οι κομμουνιστές. Μέχρι που το 1992 πέτυχε αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Κροατίας. Από τότε η Κροατία με μεταρρυθμίσεις και διαπραγματεύσεις βρίσκεται στην άγουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια χώρα της ε, κεντρικής ευρωπαϊκής Ευρώπης, μια από τις υποψήφιες χώρες καλύτερα προεδρεσμένη από οποιαδήποτε άλλη. Και θα ήθελα αγαπητέ ε, συνάδελφε Σφόβοντα να σας πω πόσο χαίρομαι ότι μπορέσαμε τους άλλους σκιώδεις και εισηγητές όλα αυτά τα χρόνια να καταφέρουμε αυτό εδώ το σώμα να είναι εκείνο που εξάλληψε κάποια άδικα εμπόδια που υπήρχαν στην, στο δρόμο της Κροατίας αυτή η χώρα τεχνητά είχε μπλοκαριστεί με απαράδεκτο τρόπο. Είναι ήδη αρκετά δύσκολη η φυσιολογική διαδικασία ένταξης, αλλά οι διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στην Κροατία ήταν οι πιο αυστηρές από ε, εκείνες που επιβλήθησαν σε οποιαδήποτε άλλη υποψήφια χώρα. Η Κροατία κατάφερε να ξεπεράσει τα αμπόδια αυτά θαυμάσια και γι' αυτό χαίρομαι που σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε παρατηρητές από την Κροατία που θα μας βοηθήσουν να δώσουμε μια νέα όθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι που θα μιλάτε ε, κροατικά. Ζήτω η Κροατία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πόσελ. Τώρα για την ομάδα ε, Δημοκρατών Σοσιαλιστών, ο κύριος Βίγγενιν για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ. Είμαι πεπισμένος ότι θα ήταν πιο επίσημη σημερινή συνεδρία εάν είχαμε δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα οικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και αν οι πολίτες της Κροατίας μπορούσαν να ακούσουν τι λένε οι συνάδελφοι, ίσως θα ξανασκεφτώσουν αν θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι. Η τη Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μεγάλη επιτυχία για τη χώρα αυτή και για την σύνολη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η Κροατία έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια ειδική και ξεχωριστή χρονική στιγμή. Αλλά αυτό μας βοηθάει να πιστέψουμε και εμείς ότι δεν είναι τόσο τραγική η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ακόμα ένα μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξακολουθούμε να είμαστε ελκυστικοί. Θα ήθελα να πω κάτι που είχε πει ένας άλλος εκπρόσωπος χώρας υποψήφιες. Λέτε ότι είναι πολύ δύσκολο να μπει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρετε όμως τι σημαίνει να είσαι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δέχεσαι τα χτυπήματα της κρίσης. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πάρει με μεγάλη ψηφοψηφία μια θετική στάση για την είσοδο της Κροατίας, όπως έκανε και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ήδη. Πιστεύω λοιπόν ότι το βασικό εγχείρημα στο οποίο πρέπει να αποδειθεί η Κροατία είναι να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη. Ξέρουμε ότι το χρονοδιάγραμμα <clears throat> της ε, κύρωσης είναι στενό, αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσει σύντομα η Κροατία να είναι μαζί μας ως χώρα μέλος. Χαίρομαι πολύ που ο κ. Σφόμποτα ως εκπρόσωπος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ήταν ε, ο συντάκτης μιας λαμπρής έκθεσης και βοήθησε με τον τρόπο αυτό την Κροατία να επιτύχει τους στόχους τους. Κάτι ακόμα που θέλω να υπογραμμίσω σε αυτή την έκθεση είναι το θέμα της συμμετοχής των πολιτών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε ότι με το δημοψήφισμα θα φανεί και η θετική στάση των πολιτών. Δηλαδή το δημοψήφισμα που θα γίνει στην Κροατία. Και τώρα για τον κύριο Πόσελτ. Η Κροατία χρειάστηκε να αντιμετωπίσει υψηλότερα προαπαιτούμενα από άλλε χώρε. Αυτό σημαίνει όμω ότι δεν χρειάζεται και μηχανισμού παρακολούθηση, όπω έπρεπε να αντιμετωπίσουν η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Καλή επιτυχία λοιπόν. Τώρα την ομάδα των ο κύριο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε και αγαπητοί προσκεκλημένοι από την Κροατία που βρίσκεστε στα, θεωρία είναι μεγάλη τιμή για μας που είσαστε εδώ για να παρακολουθήσετε αυτή την ιστορική μέρα που είναι τόσο σημαντική και για εσάς αλλά και για μας. Η Κροατία έπρεπε να περιμένει πολύ για να φτάσουμε σε αυτή την χρονική στιγμή και πιστεύουμε και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάλι χαρούμενα βλέμματα όταν υπάρξει και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πιστεύω ότι η Κροατία χρειάστηκε να εργαστεί σκληρότερα από άλλες υποψήφιες χώρες οι οποίες μπήκαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα μιας λανθασμένης αντιμετώπισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι δηλαδή η Κροατία ήταν μία από τις χώρες που ήταν υπεύθυνε για τον πόλεμο της πρώην Ιουκοσλαβίας. Ενώ στην πραγματικότητα η Κροατία είναι το μεγαλύτερο θύμα αυτής της, ε, της σύραξης Σήμερα ξέρουμε ότι το ευρωπαϊκό μέλλον της Κροατίας <clears throat> είναι κάτι το οποίο επετεύθη με τη συγκροτημένη προσπάθεια του λαού της Κροατίας και των πολιτικών της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια χώρα η οποία στην ιστορία της δεν ήταν πάντα μια χώρα με ενιαίες απόψεις και ενιαίες κατευθύνσεις. Σήμερα υπάρχει όμως η κοινή συνείδηση και θέληση όλων των πολιτών της Κροατίας να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκε σε αυτό τώρα και σε αυτήν την κοινή θέληση ο κύριο Επίτροπο και μονάχα μπορώ να επικροτήσω αυτά τα οποία λέει. Είναι πολλοί τομεί στου οποίου η Κροατία πρέπει να αναβαθμίσει την απόδοσή τη για την προστασία των μειονοτήτων, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλα αυτά. Αλλά αυτά δεν είναι μονάχα ειδικά προβλήματα τη Κροατία, αυτά είναι προβλήματα όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. <clears throat> Γι' αυτό θέλω να πω και εγώ καλώ ήλθε Κροατία και με μεγάλη χαρά θα την χαιρετήσουμε στο 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τάνοκ θα πάρει το λόγο για δύο λεπτά από τους Ευρωπαίους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Madam President, I had the pleasure of spending my summer holidays. Εγώ περνώ τα καλοκαίρια μου στην Κροατία και έχω δει το επίπεδο ευημερίας και κοινωνικής προόδου σε αυτή την εξαιρετικά όμορφη χώρα. Φυσικά και θα συμφωνήσουμε αύριο σαν πολιτική ομάδα για να γίνει η Κροατία το 28ο μέλος. Η Κροατία δείχνει το παράδειγμα στους γείτονες. Έβαλε στη φυλακή ακόμα και ένα τέος πρωθυπουργό για διαφθορά. Αυτό σημαίνει ότι πληρεί τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Υπάρχουν πολλά να γίνουν ακόμα στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και των εκτοπιμένων πληθυσμών. Συνεργάζεται πλήρως με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έτσι ώστε να μπορέσει να αφήσει πίσω το μαύρο παρελθόν της πρόσφατης ιστορίας. Είναι μια μεσογειακή χώρα, μια ευημερούσα χώρα, λίγα προβλήματα θα έχει να αντιμετωπίσει ε, θα έχει βέβαια το θέμα της προσωρινής εξαίρεσης ελεύθερης μετακίνησης των εργαζομένων, ιδιαίτερα προς χώρες οι οποίες συστηματικά υφίστανται μεταναστευτικές πιέσεις όπως η χώρα μου. Νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν ε, <clears throat> μέτρα όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των ε, Κροατών στην περιοχή Σέγγεν. Δυστυχώς υπάρχει κατάχρηση αυτών των ρυθμίσεων και πάρα πολλοί βέβαια ποινικοί θα έλεγα κυκλοφορούν ανεμπόδιστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα καλό παράδειγμα για τις γειτονικέ χώρες όπως το Μαυροβούνιο για την οποία είμαι εισηγητής και με την οποία έχει μία μεθοριακή διαφορά. Και η Μακεδονία, λέει ο μιλητής, θα ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις σύντομα. Το πότε θα γίνουν μέλη βέβαια οι άλλες χώρες είναι κάτι το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα αλλά παρόλα αυτά το παράδειγμα της Κροατίας είναι ένα σωστό παράδειγμα για τις προσπάθειές τους για τη δημοκρατία και νομίζω ότι η Κροατία με τη σειρά της θα πρέπει να υποστηρίξει τους παλαιούς περιφερειακούς τεχθρούς της στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην Ένωση και αναφέρομαι κυρίως στη Σερβία. Κύριε Πόσελτ, μπλε κάρτα. Θέλετε να κάνετε μια ερώτηση στον κύριο Τάνοκ. Σύντομα σας παρακαλώ. Κύριε Τάνοκ, δέχεστε μια ερώτηση από τον κύριο Πόσελτ. Yes, you Χαίρομαι ακούγοντα την ομιλία του συναδελφού Τάνοκ. Αλλά αναφέρθηκε στην ατέο πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν ξέρει βέβαια ότι χωρί αυτό τον πρωθυπουργό η Κροατία δεν είχε φτάσει εκεί που έφτασε σήμερα και μήπω πιστεύει δεν πιστεύει ότι αξίζει σωστή δίκη αυτός ο άνθρωπος. Δίκαιη, χωρίς μια εκ των προτέρων καταδίκη πολιτικά. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι στην δικαστική διαδικασία. Είναι σαμπιούντισε και επομένως δεν πρέπει να το σχολιάσω. Ξέρω όμως ότι ο Δόκτωρ Σάναντερ έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο για να ανοίξει το δρόμο για την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας πολύ ικανός πολιτικός, αν όμως είναι ένοχος διαφθοράς και κατάχασης θα πρέπει να πάει στη φυλακή. Αυτό είναι πολύ σαφές, αλλά αυτό πρέπει να το αποφασίσουν τα δικαστήρια και όχι το κοινοβούλιο μας. Για την απάντηση τώρα από την ομάδα των Πρασίνων, για 1,5 λεπτό ε, έχει το λόγο κυρία Λούνατσεκ. Πρόεδρε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Είναι πολύ καλές αυτές οι μέρες για την Κροατία αλλά και για τη σύνολη Ευρώπη. Και δεν είναι πολλές οι χαρούμενες τέτοιες μέρες που μπορούμε να ζούμε στην Ευρώπη τον τελευταίο καιρό. Η υπογραφή λοιπόν της συμφωνίας της, ένταξης, της συνθήκης ένταξης για την Κροατία την επόμενη εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ θετική. Θα ήθελα από την πλευρά της ομάδας των Πρασίνων και της Ελεύθερης Συμμαχίας να συγχαρώ εκ βάθους καρδίας τους με την ε, θετική ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την υπογραφή της συνθήκης ένταξης τελειώνουν 10 χρόνια προσπαθειών. Η διαδικασία όμως δεν θα έχει περατωθεί πλήρως. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν και περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπιστεί η διαφθορά, να υπάρξει μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, να υπάρξει διωγμός των εγκλημάτων, εγκλημάτων πολέμου και είναι όλα αυτά πάρα πολύ σημαντικά για τη διαδικασία της μεταρρύθμισης. Γι' αυτό Νομίζω ότι η τροπολογία του ΕΛΚ είναι τελείως λανθασμένη. Γιατί αναφέρεται, για, ε, αναφέρεται στις ε, ταραχές που έγιναν σε μία εκδήλωση λεσβιών, ομοφιλοφίλων κτλ. Όλα αυτά δείχνουν ένα είδος ε, επικίνδυνων στοιχείων αντιμετώπισης των ε, ομάδων στην κοινωνία αυτή. Είναι απαραίτητο λοιπόν η Κομισιόν να έχει μεγάλη προσοχή για τα θέματα αυτά και να εξασφαλίσει ότι και στην Κροατία υπάρχει μια απαραίτητη πειθαρχία και η σωστή διαδικασία εποπτείας και ελέγχου τα επόμενα χρόνια. Εμεί θέλουμε ό,τι κάνει η Κροατία να το κάνουμε με έναν τρόπο ο οποίο θα είναι διάφανο και να μπορέσουμε να πείσουμε του Κροάτε ότι όλα αυτά είναι προ το δικό του συμφέρον και επομένω με τον τρόπο αυτό θα δώσει μια όθηση σε όλε τι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων να συνεχίσουν μια θετική κίνηση προ την κατεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα το λόγο θα πάρει για ένα λεπτό, σεβαστείτε το χρόνο και συνάδελφο, ο κ. Χατζηγεωργίου από την Ενωτική Αριστερά. Once again. Μία ερώτηση έχω προ την ε, συνάδελφο Λούνασεκ. Εάν διάβασε το κείμενο το ΑΕΛΚ βέβαια είναι υπέρ τη καταδίκη αυτή τη βία Στο σημείο 14 είμαστε κατά του να αναφέρεται στο σημείο 15 ότι ήταν πτέσμα τη κυβέρνησης. Εκεί είμαστε αντίθετοι. Είμαστε βέβαια υπέρ της ε, καταδείξης τη ε, βία και των βιοπραγιών. Μάλιστα. Ε, βέβαια το διάβασα στην Αλφεπόσαλ και βέβαια εδώ δεν πρόκειται να υπάρχει εκλογικό αγώνα που να υποστηρίξουμε προ εδώ εκεί. αλλά νομίζω ότι πραγματικά έφταιγε η κυβέρνηση ότι δεν προστάτευσε του ανθρώπου εκεί στο σπλίτ κατά τη διάρκεια τη ε, διαδήλωση αυτή. Και γι' αυτό ελπίζουμε να αποσύρετε η τροπολογία σα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηγεωργίου. Συγγνώμη, είναι η ώρα σα τώρα. Ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά χαιρετίζουμε την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπαίνει βεβαίως σε μια εποχή όπου η πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοντεύει στον ναδύρ Μακάρι αυτό να αναζωογονήσει η ένταξή της στο βαθμό που μπορεί την πίστη ότι μαζί μπορούμε καλύτερα. Δεν είμαι αισιόδοξο και ακόμα παραπάνω ελπίζω ότι η ένταξη της Κροατίας δεν θα συμπέσει με την διάλυση του ευρώ και των ονείρων τόσων πολλών δεκαετιών η έκθεση προόδου του 2011 αναφέρει πως η ενταξιακή πορεία έχει δώσει στην Κροατία όθηση για θετικές αλλαγές με αποτέλεσμα να σημειώσει ουσιαστική πρόοδο σε διάφορους τομείς. Θέλουμε και εμείς να χαιρετήσουμε την πρόοδο που έχει γίνει στον τομέα της επιστροφής των προσφύγων, της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των διακρίσεων καθώς και στη γεφύρωση των διαφορών με τις γειτονιάζουσες χώρες. Πέρα όμως από αυτά θα πρέπει να μεριμνήσουμε και για τα σημαντικότερα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν τον λαό της Κροατίας, όπως η φτώχεια, η μακροχρόνια ανεργία και η καταπάτηση εργατικών δικαιωμάτων. Δυστυχώς οι προτάσεις για προώθηση μιας ανταγωνιστικής φιλελεύθερης οικονομίας θα επιβαρύνουν την ήδη δύσκολη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση του λαού. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε την προώθηση μιας πραγματικής κοινωνικής ανάπτυξης μέσω του εξυγχρονισμού του συστήματος κοινωνικής προστασίας με φιλολαϊκά μέτρα για αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων και της ανεργίας και για βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες ιδιαίτερα της υγείας, της στέγασης και της ε, εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φέρετς από την ε, ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας Δημοκρατίας για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πήγα πρόσφατα στην Κροατία, ήθελα να δω αν υπήρχε πραγματική εθνική συζήτηση, αν υπήρξε κάποια εκστρατεία για όλα αυτά τα θέματα. Τι βρήκα, βρήκα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ό,τι μπορεί για να χρηματοδοτήσει για να χρηματίσει την πολιτική ελίτ της Κροατίας. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει 320 εκατομμύρια στην Κροατία σε προενταξιακή βοήθεια όπως λέγεται και έχει εξοδέψει ένα εκατομμύριο για χτυπητή εκστρατεία προπαγάνδας λέγοντας στους Κροάτες τι καλύπτουν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως δώσατε και δουλειές καλοπληρωμένες δουλειές σε Κροάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν για να τους δείξετε τι ωραία που θα περνάνε οι κυρίαρχες τάξεις αν μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναπετάνονται οι σημαίε της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε, στη κεντρικά κτίρια της πρωτεύουσα για να φανεί ότι έχει τελειώσει αυτό το πράγμα και είναι δεδομένη η ένταξη. Αλλά έχουμε ακόμα μία ελίτ που κρατάει την εξουσία στην Κροατία είναι αυτοί που θα υποφεληθούν οικονομικά από την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και μια ακόμα πιο αρνητική και σκοτεινή πλευρά. Δεν υπάρχει ελεύθερος τύπος στην Κροατία. Δεν υπάρχει καμία εθνική συζήτηση που να λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή. Έχει δοθεί ένα βραβείο 10.000 κονών για οποιονδήποτε μπορεί να βρει ένα άρθρο σε μια εφημερίδα της Κροατίας που να λέει κάτι εναντίον της ένταξης. Όλη αυτή η διαδικασία είναι στρεβλή και διεφθαρμένη και βλέπουμε να γίνεται κάτι που έχει γίνει και στο παρελθόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα στην Κροατία. Η χώρα αυτή διεκδικεί την ανεξαρτησία της εδώ και χίλια χρόνια. Για 20 χρόνια είχε την ανεξαρτησία της, βγήκε από το λανθασμένο πολιτικό πείραμα της Ιουκοσλαβίας, αλλά τώρα αν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπει σε μια νέα Ιουκοσλαβία, Ιουκοσλαβία μεγάλη μεγαλύτερη, ένα μεγαλύτερο αποτυχημένο πολιτικό πείραμα. Δυστυχώς δεν δε βλέπω να γίνεται συζήτηση για αυτό το θέμα στην Κροατία. Τώρα ο κύριος Μπρόνς από τους μη εγγεγραμμένους για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κύριος Μπρόνς. Uh, Εδώ και 20 χρόνια διακήρυξε την ανεξαρτησία της μετά από ένα δημοψήφισμα με 95% υπέρ της ανεξαρτησίας και του λαού της. Πόλεμος έγινε τότε, πολλοί σκοτώθηκαν για να υπερασπιστούν τα εθνικά τους συμφέροντα και είναι τραγικό ότι στην ουσία παραδίδει την ανεξαρτησία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να επιβάλλει νομοθετικές ρυθμίσεις κοινωνικού τύπου και να δημιουργήσει γενικά καταστάσεις απαράδεκτες και να προσυπογράψει έναν οικονομικό φιλελευθερισμό ο οποίος θα υπονομεύσει τα συμφέροντα του λαού της χώρας. Όλα αυτά δείχνουν περιφρόνηση της δημοκρατίας, περιφρόνηση του κροατικού λαού και περιφρόνηση των νεκρών της Κροατίας στον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Η κυβέρνηση της Κροατίας όχι μόνο έχει χρησιμοποιήσει καταχρηστικά το δημόσιο χρήμα για την προπαγάνδα υπέρ του δημοψηφίσματος, αλλά αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος σαν κάτι το εντελώς τυπικό αν δεν υπάρξει θετική ψήφος έτσι κι αλλιώς τη σημασία έχει θα γίνει κι άλλο δημοψήφισμα και μετά κι άλλο ώσπου να μάθουν και να ψηφίσουν θετικά. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, κυρίες και κύριοι, η διαδικασία λήψης απόφασης κατέδειξε, θα το δούμε αύριο, ότι πρόκειται για καλές μέρες, όχι μόνο για την Κροατία, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση με την απόφαση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν το σχέδιο της Ένωσης της Υπήρου, σαν το σχέδιο της υπέρβασης της βίας, ε, του διαχωρισμού της Ευρώπης, σαν ένα σχέδιο της ευθύνης για αλλήλους και όχι της, ε, του πολέμου των μεν αντίον των δε. Υπέρβαση της κρίσης και η αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας. Η διαδικασία διεύρυνση δεν έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία εμβάθυνση πρέπει να επιτεχυνθεί. Η κοινωνική και η οικονομική ένωση πρέπει να ιδρυθεί, πρέπει να τελειοποιηθεί. πρέπει να δράσουμε σωστά. Και στην Κροατία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να επαναπαυθούμε στις δάφνες ε, μας, θα πρέπει να συνεχίσουμε στην οδό των μεταρρυθμίσεων και στην Κροατία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης, καταπολέμηση διαφθοράς και προάσπιση των βασικών δικαιωμάτων και προώθηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι ο συνάλφος και η κυρία Λούνασεκ, ο υποφαινόμενος και ο κύριος Πόσελτ εδώ και χρόνια παρακολουθούμε την άγουσα αυτή. Η Αυστρία είναι μετά αξία εκείνων των χωρών που πρώτες αναγνώρισαν την εξαρτησία της Κροατίας. Οικονομικά, όσον αφορά την απασχόληση, πολιτιστικά, ιστορικά, είμαστε ενωμένοι με τη χώρα αυτή και γι' αυτό χαιρόμαστε που η διαδικασία αυτών των τελευταίων ετών μπόρεσε να ολοκληρωθεί επιτυχώς. Και ελπίζουμε όλοι αύριο να πούμε ένα ξεκάθαρο ναι και εγκάρδιο καλαθοσόρισμα προς την Κροατία και από κοινού να δώσουμε τις απαραίτητες οθήσεις που χρειάζεται για να προχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Οδό από κοινού. Και η εικόνα και για τα δικά είναι θετική. Κάρας. Τώρα η κυρία Φαγιόν για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κυρία Φαγιόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η υποστήριξη της Κροατίας αύριο θα είναι ένα σημαντικό σημάδι από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι ακόμα και στις δύσκολες αυτές στιγμές η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να προχωρά. Και θα είναι και ένα πολύ καλό μήνυμα για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων η είσοδο τη Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντική για όλε τι χώρε τη περιοχή, γιατί η Κροατία μπορεί να είναι το θετικό παράδειγμα για άλλε χώρε τη περιοχή που πρέπει να λύσουν τα μεταξύ του προβλήματα και με τον τρόπο αυτό μπορούν να εξασφαλίσουν ένα καθεστώ αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ του. Το αποτέλεσμα τη διαμεσολάβησης μεταξύ τη ε, Κροατία και τη Σλοβενία ήταν θετικό. Η Κροατία επίσης προχώρησε σε πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και αυτές οι μαραθώνιες προσπάθειες αλλά και το τελικό σπριντ θα πρέπει να ευοδοθούν και να ανταμυφθούν. Οι πολιτικοί λοιπόν πολλές φορές κάνουν λάθη και αλλάζουν την ισορροπία που πρέπει να υπάρχει στην περιοχή των Βαλκανίων. Αλλά είναι ο λαός ο οποίος πρέπει να αποφασίσει αν θέλει πράγματι να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι και στην Κροατία, όπως και στη Σλοβενία στο παρελθόν, θα είναι θετικό το δημοψήφισμα και αυτό θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα στην περιοχή της Κροατίας και θέλω να συγχαρώ και να χαλωσορίσω τους συναδέλφους από την Κροατία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ο κύριος Βόμποντα είναι σοβαρός άνθρωπος και μας έχει φέρει μια άρτια και σοβαρή έκθεση. Πρέπει όμως να τονίσω ότι έχει κάνει σοβαρές προσπάθειες και η Κροατία για να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε. Έτσι έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς και υπολογίζω να συνεχίσει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για την ίδια, με την ίδια δυναμική, ειδικότερα όσον αφορά τους τομείς της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τις βελτιώσεις στον εγχειρισμό των υποθέσεων διαφθοράς, την δημόσια διαφάνεια στον τομέα των προμηθειών, την χρηματοδότηση των κομμάτων. Σε αντίθεση με άλλα υποψήφια κράτη της περιοχής, έχει παρουσιάσει μια τεράστια πρόοδο και αναφέρομαι στη ΦΥΡΟΜ η οποία υπολείπεται και ανεξαρτήτως του ονόματος δεν είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διαδικασίες. με την έννοια αυτή σε κάθε περίπτωση ελπίζω ότι η ένταξη της κροατίας θα δώσει νέα πνοή στην ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των δυτικών βαλκανίων και με αυτή τη φράση καλωσορίζω την κροατία στην ευρωπαϊκή ένωση. ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενο ομιλητή εγγεγραμμένο είναι ο κύριο Κόβατ. Δεν φαίνεται να είναι στην αίθουσα. Και θα δώσω στον κύριο Χόκμαρκ τον λόγο για δύο λεπτά. Μίστερ Χόκμαρκ. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Two minutes, please. Χωρίς μικρόφωνο μιλητής. Micro, please. Thank you. Madam Speaker, I would like to thank the... Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Θέλω να καλωσορίσω την Κροατία και να συγχαρώ Κλείνει το μικροφόνο το μιλητής δυστυχώς. Κάποιος μου κάνει σαμποτάζ εδώ. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να ψηφίσουμε για την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα είναι και μία εκδήλωση και απόδειξη της επιτυχίας της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Λυπάμαι που έφυγε ο κύριος Φάρατς γιατί είχε ένα πρόβλημα με την ένταξη της Κροατίας. Γιατί η ένταξη της Κροατίας είναι ένα μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αξίες οι οποίες είναι πιο ελκυστικές από τις δικές του ιδέες. Και καταδεικνύει ότι σε καιρούς κρίσης μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει ένα από τα θαυμάσια εγχειρήματά της, με την διεύνηση. Όλα αυτά τα οποία είδαμε είναι ότι έχει έλθει η σταθερή δημοκρατία σε πολλές κοινωνίες της Ευρώπης. Και χάρη στην Κροατία θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο πέρα και να κάνουμε ακόμα καλύτερα, καλύτερη την Ευρώπη. Έχει γίνει καλύτερη κοινωνία η Κροατία. Οι πολίτες της θα έχουν όλες τις ευκαιρίες που έχουν οι υπόλοιποι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα κάνει και καλύτερη την Ευρώπη αυτή η ένταξη. Θα δημιουργήσει καλύτερες ευκαιρίες για όλους μας. Όλοι αυτοί οι πολίτες της Ευρώπης, είτε από την Κροατία, από τη Σουηδία, από την Αυστρία, από κάπου αλλού, θα έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο να καταδείξουν την αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καιρό οικονομικής κρίσης. Και έτσι θα έχουμε καταδείξει ότι υπάρχει χώρος για αισιοδοξία και υπάρχει περιθώριο για ένα θετικό μήνυμα προς άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Αν αλλάξετε, αν μεταμορφωθείτε, αν αναπτυχθείτε, μπορούμε όλοι από κοινού να ζήσουμε σε μια δημοκρατική, ανοιχτή κοινωνία και ευ ευμαρή κοινωνία. Για 1,5 λεπτό φυσικά και θα υπερψηφίσουμε την ένταξη της κροατίας. Είμαι από μια γειτονική χώρα, θέλω να συγχαρώ λοιπόν δύο φορές τη χώρα αυτή. Είναι παράδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής που θέλουν και αυτές να γίνουν μέλη. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι ότι είναι εφικτό να γίνει κανείς μέλος και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Έκλεισαν τα τελευταία κεφάλαια και κατά τη διάρκεια της τελευταίας Ουγγρικής Προεδρίας πάντα ήμασταν υπέρ της Κροατική υποψηφιότητα Υπάρχουν κάποια βήματα που πρέπει να κάνει ακόμα βέβαια η Κροατία και το λέγω αυτό από μια χώρα η οποία σχετικά πρόσφατα έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καλό το να προωθεί κανείς ε, καλές σχέσεις γειτονίας, το να θέτει τέλος σε μια παράδεκτη μερικές φορές εθνικιστική ρητορική, ιδιαίτερα στα πλαίσια αυτής της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε τις τόσο σοβαρής. Εμείς θα πρέπει να προωθήσουμε τις αξίες μας και με την κυβέρνηση της χώρας και με όλους τους, κοινο... τους συναδέλφους της Κροατίας να ενημερώσουμε σωστά τους πολίτες τι σημαίνει να είναι κανείς ε, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο επόμενος εγγεγραμμένος ομιλητής δεν είναι στην αίθουσα και θα δώσω το λόγο στον κύριο Πέτερλε για ένα λεπτό παρακαλώ. Euh, euh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ την Κροατία για την περάτωση των διαπραγματεύσεων και την προσεχή υπογραφή της συμφωνίας της συνθήκης ένταξης. Καταδεικνύει λοιπόν αυτό ότι έχουμε καταφέρει να προωθήσουμε τη διαδικασία διεύρυνσης και ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η δεύτερη χώρα από την περιοχή της πρώην Ιουκοσλαβίας που γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω και ελπίζω ότι αυτό θα οδηγήσει και άλλα κράτη τη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία και να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό θα αυξήσει την σταθερότητα, την ειρήνη και την συνεργασία στην περιοχή αυτή. Το λόγο για ένα λεπτό όπως είχε προβλεφθεί. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο παρόλο που προηγουμένως αποσίαζα. Ε, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και θα ήθελα να υποστηρίξω όλους τους ότι η Κροατία πραγματικά είναι η χώρα που είναι καλύτερα από οποιαδήποτε προετοιμασμένη για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δύο τελευταίου μήνε ε, επετέχθησαν πολλέ βελτιώσει και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Ένωση και του ε, εταίρου μα στην Κροατία για τι προσπάθειε που κατεβλήθησαν. Το θέμα είναι ότι έχουμε σαφεί κανόνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιοι είναι οι όροι που πρέπει να τηρεί μία χρόνια. Και αυτό που με λυπεί είναι ότι δυστυχώ πάλι δεχόμαστε μία χώρα η οποία δεν πληρεί 100% τις προϋποθέσεις. Εγώ δεν θέλω να υπάρχουν μειονεκτήματα, να είμαστε αρνητικοί εναντί της Κροατίας. Έχει προχωρήσει από οποιοδήποτε άλλη, αλλά θα ήθελα στο μέλλον να υπάρχει ισότητα στο δίκαιο και όχι στο άδικο. Γιατί πραγματικά έχουμε εδώ καλούς κανόνες και γι' αυτό είμαστε τόσο ελκυστικοί. Θα είναι άσχημο όταν δεν τηρούμε τους κανόνες και θα ήθελα να τηρηθούν στην επόμενη διάβριση. Ευχαριστώ κύριε Κάσπαρη. Τώρα, ε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ερχόμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχουν ζητήσει αρκετοί συνάδελφοι το λόγο. Θα τον πάρουν μόνο έξι. Ξεκινάω από τον κύριο Μίκολα Σίκ. Κρατήστε το χρόνο του ενός λεπτού για να μπορέσουν να μιλήσουν και οι έξι, αντί για πέντε που, που ήθιστε. Κύριε Μικολασίκ, ένα λεπτό παρακαλώ. Δεν είναι στην αίθουσα. Μίστερ Μικολασίκ. Λοιπόν, δεν τον βλέπω. Η κυρία Ρότοβα, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η επιτυχής ολοκλήρωση των διαδικασιών της Κροατίας είναι κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Η Κροατία είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Ταυτόχρονα είναι και μια εγγύηση θα έλεγα για τη σταθερότητα της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων. Είχαμε πάρα πολύ στενές σχέσεις με την Κροατία, ενώ ανάμεσα στην Τσεχία και στην Κροατία. Α, και από την άλλη Βλέπω ότι η τσεχική ε, διαδικασία περιπλέκει ε, την υποψηφιότητα της Κροατίας λόγω ακριβώς των ε, πολιτικών θεμάτων που έχει θέσει η σοσιαλδημοκρατία στη χώρα μου, στην Τσεχία. Όλα αυτά όμως δεν πρέπει να καθυστερήσουν την ένταξη της Κροατίας. Με το συμπληρωματικό πρωτόκολλο το οποίο θέλει να υπογραφεί η Τσεχία περιπλέκει την κατάσταση Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να διευκολύνουμε τις διαδικασίες της Κροατίας. Συγχαρητήρια και τον Επίτροπο Φούλε. Παρακαλώ. Τώρα ο κύριος Κασίν έχει το λόγο. Παρακαλώ, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πάλι οι ευρωσκεπτικοί εθνικιστές παίρνουν κακό βαθμό. Θέλω γι' αυτό να συγχαρώ την Κροατία και επίσης και την Πολωνική Προεδρία. Θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι περήφανοι για το σημαντικό αυτό επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ευχαριστήσω και τον Χάνης Σφόμποτα για τη μακροχρόνια και θετική του εργασία. Στις 19 Δεκεμβρίου θα πρέπει να παραδώσουμε τη σκητάλη και να ορίσουμε μία ημερομηνία συγκεκριμένη για την Κροατία. Η Κροατία αξίζει την ένταξή της και η Ευρωπαϊκή Ένωση αξίζει τη νέα αυτή χώρα. Θα πρέπει να την υποστηρίξουμε λοιπόν στις προσπάθειες αυτές και θα ήθελα να παρακαλέσω την Πολωνική Προεδρία καθώς επίσης και όλο το Συμβούλιο και την Κομισιόν εκτός από την Κροατία να προσθέσει το Μαυροβουλίο και τη Σερβία. Κυρία Τσικάου, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι με το γεγονός αυτό θα υπάρξει μια σημαντική συνεισφορά για να εφαρμοστεί η στατική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη. Ξέρουμε ότι η Κροατία με την Γερμανία είναι υπεύθυνε για τον άξονα υπεριθμών 6 για την προστασία της βιοπικιλότητος στην περιοχή αυτή. Η Ρουμανία είναι αρμόδια για τον άξονα 8, ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η Κροατία λοιπόν σαν κάτω μέρος μπορεί να βοηθήσει να υπάρξει καλύτερη ε, ανάπτυξη των ε, διευρωπαϊκών δικτύων. Η Κροατία λοιπόν μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την διεύρυνση των υποδομών της Ευρώπης σε επίπεδο συγκοινωνιών και να υπάρξει και περάτωση στην περιοχή των Βαλκανίων. Παρακαλώ, κύριος Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μετά από πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια, ευτυχώς θετικά ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσει έναξη τη Κρατίας. Αυτό πρέπει να το χαιρετήσουμε γιατί πολλά έγιναν στην Κροατία τα μεταρρύθμιση δικαιοσύνη Φερρυπίν. Από την άλλη μεριά είναι αναγκασμένη η Κροατία να συνεχιστεί να σκέφτεται το θέμα της ε, εξόδου από την πυρηνική ενέργεια και της, ε, του κλεισίματος ορισμένων πυρηνικών σταθμών. Επίσης, πολέμηση διαφθοράς, ε, ανθρώπινα δικαιώματα, ανταγωνισμός, όλα αυτά είναι θέματα σημαντικά η Κομισιόν πολλά ζήτησε από την Κροατία, πολύ περισσότερα από οποιασδήποτε άλλες υποψήφιες χώρες. Και η Κροατία μπόρεσε να ε, προχωρήσει και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Τουρκία δίνουν δισεκατομμύρια για το Βόσπορο. Πού κάνει για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η ψηφοφορία που θα γίνει αύριο για την ένταξη της Κροατίας είναι ένα πραγματικό και σημαντικό ορόσημο για μας. Νομίζω ότι θα ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση η ένταξη της Κροατίας και θα αυξήσει και την αξιοπιστία της. Η διαδικασία ένταξης έχει οδηγήσει σε μια μεταμόρφωση της ε, Κροατίας και είμαι πεπισμένος ότι με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η σταθερότητα, η ασφάλεια και η ελευθερία στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Η Κροατία εκπροσωπεί λοιπόν τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές και θα είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε και τις άλλες χώρες της περιοχής που θα πρέπει να ακολουθήσουν και θα πρέπει να εστιάσουμε τις κοινέ μας προσπάθειες ως Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατεύθυνση αυτή. Η επιτυχία λοιπόν της Κροατίας θα είναι ένα δίδαγμα και ένα υπόδειγμα και για άλλες χώρες της περιοχής. Θέλω λοιπόν να χαιρετήσω ιδιαίτερα την Κροατία ως 28 ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Az Európai Unió jelenleg talán történelme legnehezebb időszakát éli, amikor az Αυτή τη στιγμή η Κροατία περνάει μια, η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της όταν η αλληλεγγύη και η εμπιστοσύνη αντικαθίστανται από εγωιστικές συμπεριφορές. Είναι απαραίτητο λοιπόν είναι το Συμβούλιο και η Κομισιόν να παραμείνουν προσιλωμένοι στην ένταξη της Κροατίας ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Δεν μπορεί να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της Ευρώπης χωρίς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Με τις χώρες αυτές είναι απαραίτητο όμως να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα των ενδογενών εθνοτικών μειονοτήτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Η ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων δεν μπορεί να γίνει αν παραγνωρίσουμε το θέμα των μειονοτήτων. Ελπίζω και πιστεύω ότι η Κροατία θα ακολουθήσει θα τηρήσει μάλλον τις υποσχέσεις της πριν από την ένταξη για την προστασία των μειονοτήτων. Ευχαριστώ. Βάστο των συναδέλφων, το λόγο θα πάρει ο Επίτροπος. Κύριε Φούλε, έχετε το λόγο. Mr. Commissioner, you Thank you very much. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, ευχαριστώ για τη συζήτηση που προηγήθηκε. Πολύ θετική συζήτηση με ενέπνευσε και με ενεθάρρυνε η υποστήριξη προς την Κροατία αύριο θα μετατραπεί σε αποφασιστική θετική ψήφο. Πράγματι η Κροατία χρειάζεται την ενθάρρυνσή σας για να συνεχίσει την προετοιμασία σας. Η έκθεση, η φθινοπορεινή την οποία προετοιμάσαμε, δείχνει ότι η Κροατία συνεχίζει την προσπάθεια και είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες του να είναι κανείς μέλος της Ένωσης. Αυτές είναι οι βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης που θα σχηματιστεί μετά τις επόμενες εκλογές. Το λέω αυτό για να υπογραμμίσω ότι δεν θα υπάρξουν φυσικά εξαιρέσεις για την Κροατία ή για οποιαδήποτε άλλη χώρα, οι στόχοι τους οποίους διαπραγματευτήκαμε με την Κροατία παραμένουν σταθεροί και η διαδικασία θα ακολουθηθεί χρονικά όπως αυτό έγινε μέχρι τώρα. Η ένταξη και η συνθήκη επί τη βάση του άρθρου 49 θα είναι μια συγκεκριμένη ένταξη και θα αφορά μόνο τη συγκεκριμένη χώρα. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας στη στενή με την Κροατία και θα ενημερώσουμε και το Κοινοβούλιο για την πρόοδο την οποία θα επιτελεί η χώρα αυτή τους επόμενους μήνες πριν από την ένταξη. Νομίζω ότι η πολιτική διεύρυνση είναι η απάντησή μας στην φιλοδοξία και την προσδοκία των λαών της Ευρώπης να συνεργαστούν ακόμα στενότερα και νομίζω ότι πράγματι το παράδειγμα που ακολουθήθηκε στην περίπτωση της Κροατίας δείχνει ότι η πολιτική μας είναι μια σωστή πολιτική. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Νταουγκίλεβιτς από πλευράς του Συμβουλίου. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε, αγαπητά μέλη. Και εγώ θέλω να χαιρετήσω και την κροατική αντιπροσωπεία στα θεωρία. Να τους συγχαρώ για την πολύ καλή και σκληρή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια που οδήγησαν την Κροατία στην πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και νομίζω ότι όταν μπουν και οι Κροάτες θα συνηθίσετε και εσείς όλοι οι υπόλοιποι περισσότερο τα σλαβικά ονόματα όπως το δικό μου που σας φαίνεται πολύ δύσκολο, Νταουγκίλεβιτς Να πω ότι ενθυμούμε πολύ καλά όταν το Κοινοβούλιο είχε ψηφίσει στο Στρασβούργο το 2003 την ένταξη όλων των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Θυμάμαι τις συζητήσεις που είχαν γίνει και πριν από τα δημοψηφίσματα που έγιναν σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και στη δική μου χώρα, και ακούσαμε και αρκετές ευρωσκεπτικιστικές ανοησίες οι οποίες κυκλοφορούσαν τότε από παντού σχετικά με την οικονομική καταστροφή η οποία θα ακολουθούσε, το τέλος της γεωργίας, το τέλος του χριστιανισμού, το τέλος των ηθικών αξιών, ανοησίες. Κοιτάξτε πώς πάει η Πολωνία, πόσο καλά, πάει, πόσο καλά πάνε οι χώρες της Βαλτικής. Τη σωστή συνεργασία έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι τεράστια επιτυχία ήταν η πολιτική διεύρυνση και ιδιαίτερα ο τελευταίος γύρος. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα είναι μια συζήτηση με συγκεκριμένα δεδομένα, θα βασίζεται στα πραγματικά ερωτήματα, στα πραγματικά και ουσιώδη θέματα και δεν θα επαναληφθεί η ίδια συζήτηση η οποία ήταν τυφλή και άγωνη. Πολύ μακράν από την πραγματικότητα. Αύριο λοιπόν ελπίζω να είναι θετική η ψήφος. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σβόμποντα για όλες τις προσπάθειες τις οποίες έκανε για να διατυπώσει μια σωστή έκθεση για την Κροατία. Ελπίζω, λέει ο κύριος υπουργό, ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε θα σταθούμε ικανοί να στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξία, δυναμισμού, θετικής ενέργειας που οδηγεί στην ένταξη της Κροατίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ο... Θέλω να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Σφόμποντα για την εκθέση αυτή και προσβλέπουμε στη